πορεία θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Ερχόμαστε στην τελευταία έκθεση για την στρατηγική της ψηφιακή ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική. Η συγγήτρια έχει τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Η έκθεση αυτή απευθύνεται στην ύπατη εκπρόσωπο κυρία και την εξωτερική υπηρεσία της. Οι τεχνικές εξελίξεις επηρεάζουν τη ζωή του των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο παραστατικό τρόπο. Πολλά κράτη-μέλη και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη πρόσβασης στο ίντερνετ και αυτό περιλαμβάνεται και στα κριτήρια της Κοπενχάγης. Η προώθηση, η προώθηση διαφόρων προγραμμάτων είναι ευπρόσδεκτα, αλλά πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Αύριο θα ψηφίσουμε για την πρώτη στρατηγική και δεν, δεν προτείνω υπερβολική ρύθμιση, αλλά σε ορισμένους τομείς πολιτικής πρέπει να επικαιροποιηθούν οι κανόνες βεβαίως και αυτό που να γίνεται με την κατάλληλη δημοκρατική εποπτεία. Η, περιμένει το σχέδιο της Επιτροπής με ανυπομονησία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να ε, εστιαστούμε στους ανθρώπους. Ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικός. Η χρήση του ίντερνετ, η χρήση του ίντερνετ αυξάνεται διαρκώς. Οι άνθρωποι που βρίσκονται υπό καταπίεση χρειάζονται ενημέρωση, πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημαίνει επίσης να επιτρέπουν στους ανθρώπους να αποφεύγουν την ε, λογοκρισία και τις ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Χρειάζονται βεβαίως ε, να εφαρμόζονται ποινές, χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη υψηλότερη λογοδοσία οι τεχνολογίες αυτές είναι σημαντικές, πρέπει όμως να βρίσκονται υπό έλεγχο και πρέπει χωρίς την και διότι αλλιώ υπάρχει κίνδυνο η όλη προσπάθεια εφόσον δεν στηρίζεται στο κράτος δικαίου να αποτύχει. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται για να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις κατάλληλε υποδομές ώστε να έχουν όλη πρόσβαση στη γνώση και στην ενημέρωση ακόμα και στι πιο απομακρυσμένε περιοχές. Μετά από τα ατυχήματα ε, που συνέβησαν πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνδέσεις και η ε, τεχνολογία της επικοινωνίας και της πληροφόρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρέπει να επαγρυπνούμε και να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να προωθήσουμε ή να προσπίσουμε τις ψηφιακές ε, εφαρμογές στον κόσμο εάν δεν είμαστε θέση να προστατεύουμε τις ψηφιακές εφαρμογές στις δικές μας χώρες. Πρέπει να προωθήσουμε την αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η, εξωτερική, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης προωθεί, προωθεί τις ψηφιακές ελευθερίες. Αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τα ε, πρότυπα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αναβαθμίσουμε τους νόμους μας ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής ελευθερίας. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να τα κάνουν μόνες τους. Ο ιδιωτικός τομέας έχει μεγάλες ευθύνες. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσει μόνο αν συμπεριλαμβάνει όλους μεταξύ των οποίων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και του χρήστες του ίντερνετ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το δημόσιο συμφέρον καθώς προωθούμε και προβάλλουμε το ίντερνετ το οποίο και εκείνο με τη σειρά του πρέπει να, να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον αυτή η έκθεση μας θυμίζει πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ανοιχτής και επικοινωνίας ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Τσικάου έχει το λόγο. Η στρατηγική για τις ψηφιακές ελευθερίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλά για ανοιχτά δίκτυα, ανοιχτό διαδίκτυο και ούτω καθεξής. Αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η τεχνολογία πληροφόρησης και επικοινωνίας έχει μεγάλη σημασία για την εκπαίδευση, κατάρτιση, ε, παρατήρηση εκλογών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι σωστές ε, πολιτικές, ιδιαίτερα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβάλλουν ε, μία συντονισμένη αντιμετώπιση για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στη γνώση και, στη... και ιδιαίτερα στην ψηφιακή θα πρέπει να προωθηθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προωθήσουμε τις ψηφιακές ελευθερίες ιδιαίτερα στις νέες δημοκρατίες ή σε χώρες που γνωρίζουν μια μεταβατική περίοδο. Ευχαριστούμε κυρία Τσικά, ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά την εισηγήτρια. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τις ε, ψηφιακές ελευθερίες. Έχει σημασία όμως για ποιες ελευθερίες μιλάμε. Ιδιαίτερα με τη μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου. Πρόσφατα είδαμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Είναι καλό το ότι αναγνωρίζεται ως βασικό δικαίωμα από τους ε, ανθρώπους, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τρομοκρατικές ενέργειες, τον εκφοβισμό μέσω διαδικτύου και τον έλεγχο των ολοκληρωτικών καθεστώτων που ελέγχουν τους ε, πολίτες τους. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο για να εξασφαλίσει στις, ε, τις ψηφιακές ελευθερίες στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η ψηφιακή ελευθερία είναι ένας τρόπος για να διαδώσει κανείς πληροφορίες, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τα κλειστά καθιστώτα. Αυτό σημαίνει μια περιπλοκή στον έλεγχο της κοινωνίας. Γι' αυτό αναμένουμε πως τέτοια καθεστώτα θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την ψηφιακή ελευθερία και να ελέγξουν τη ροή πληροφοριών για να μπορέσουν να ελέγξουν την πληροφορία που κυβερνούν. Ε, δεν έχω ψευδεστήσει ε, πως μέσω τεχνολογικών εμπάργων θα μπορέσουμε, εμπάργο θα μπορέσουμε παραδείγματο χάρη να εμποδίσουμε την Κίνα από το να εφαρμόσει την πολιτική της ε, στο διαδίκτυο. Θεωρώ πως στην εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να φροντίσουμε να πείσουμε αυτά τα καθεστώτα πως η κοινωνία θα αναπτυχθεί ελεύθερα και με τον ε, τρόπο αυτό και η κινέζικη κοινωνία θα είναι πιο ελεύθερη και πιο ασφαλής. Οκληρώθηκε η διαδικασία του Catch Δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση της εισηγήτριας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μπορώ να εκτιμήσω λόγω της προϋπηρεσίας μου σε άλλο τομέα στη χώρα μου τη σημασία αυτής της έκθεσης η οποία συμβάλλει στις προσπάθειες της Ένωσης για τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη, την διακυβέρνηση του ίντερνετ, το εμπόριο και την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιώντας το δεσμό όπως είδαμε στην Αραβική Άνοιξη ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως σημαντικούς τομείς για την πρόσθεση δημοκρατίας. Συμμεριζόμαστε την άποψη του Κοινοβουλίου διότι η χρήση του ίντερνετ, των κινητών τηλεφώνων και η τεχνολογία της πληροφόρησης και της επικοινωνίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτρέποντας την ελεύθερη άσκησή τους στην αναζήτηση μεγαλύτερης, περισσότερης δικαιοσύνης όπως είδαμε στη Βόρεια Αφρική παρόλα τα ε, γεγονότα τα οποία ε, οδήγησαν σε παρεμπόδιση της χρήσης του ίντερνετ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθεί να στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα σε απάντηση στην αύξηση της λογοκρισίας στο διαδίκτυο. Στην Τρίτη Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του περασμένου Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Εθνών, ή μάλλον της 6 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατήγγειλε τη χρήση λογοκρισίας στο ίντερνετ το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει στο σχέδιο δράσης του δράσεις για την ε, προώθηση διαφόρων ε, στρατηγικών Όπω, παραδείγματο χάρη η στρατηγική τη μη αποσύνδεση, εξασφαλίζοντα ότι το ίντερνετ θα παραμείνει όχημα προώθηση τη ελευθερία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, έχουν προβλεφθεί κυρώσει για την εξαγωγή αυτών των τεχνολογιών στο Ιράν και τη Συρία ώστε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να ε, ε, στραφούν εναντίον των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεχίζουν συζητήσει για την αναθεώρηση Τη του πολιτικής εξωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τη δυνατότητα να εξηγείται εξωτερικός έλεγχος πάνω σε κάποια ε, υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του διαδικτύου ή την, της, ε, των τηλεπικοινωνιών σε παραβίαση σημαντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στο φόρουμ που έγινε στον Μπάχου η, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέλη του Κοινοβουλίου ενωμένα προάσπισε την αρχή ότι περιορισμοί στις θεμελιώδεις τις ελευθερίες οποιασδήποτε μορφής και όπου λαμβάνουν χώρα είναι κάτι το απαράδεκτο ε, μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέλη Απριλίου του χρόνου θα εκδώσουμε σαφείς οδηγίες για τις, για τις εταιρείες, τηλεπικοινωνιακές εταιρείες σε ό,τι αφορά την υποχρέωση και την ευθύνη που έχουν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που, έχει θεσπίσει, ε, που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη που ονομάζονται αρχές ΡΑΚΙ. Οι εμπορικές μας συμφωνίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Υπηρεσίε Επιτροπή είναι αποφασισμένε να προ, προστατεύσουν την ψηφιακή ελευθερία σε όλε τι εξωτερικέ δράσει Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκδώσουν και μία ανακοίνωση για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Στην επικείμενη διάσκεψη για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει προσπάθειέ τη ώστε να συμμετέχει σε οργανισμούς όπως είναι ο ΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη με σκοπό να προωθήσει και να εξασφαλίσει την ε, απόλυτη ελευθερία στη χρήση του ίντερνετ. Πρέπει να δώσει το παράδειγμα εφαρμόζοντας τις πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύοντας, προωθώντας διάφορα έργα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τέλος, κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να παίξει αποφασιστικό ρόλο για την προστασία ενός κατάλληλου ίντερνετ που θα εξακολουθεί να προωθεί την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα και στα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, εξασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξή τους. Έληξη η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Σας εύχομαι σε όλους καλό βράδυ.